Θα ήθελα να χαιρετήσω τον Πρόεδρο και τον Επίτροπο. Παρακαλώ καθίστε. Έχουμε ψηφοφορία στις 5. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να σεβαστούμε το χρονοδιάγραμμα. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι μια κοινή συζήτηση που αφορά την απαλλαγή 2017. Για τη συζήτηση αυτή έχουμε 53 εκθέσεις στο σύνολό τους από 6 εισηγητές. Την κυρία Γιάλα Σέντερ, τον κύριο βάλι, την κυρία Σμιτ, τον κύριο Κον, τον κύριο Σαβάρμα και την κυρία Τεμπάλοβα. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Λένε, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ελεκτικού Συνεδρίου. Χαιρόμαστε που είστε εδώ μαζί μας και λεχθέντων αυτών. Μπορούμε τώρα να δούμε την έγκριση των πρακτικών. τα πρακτικά και το κείμενο που έχουν υιοθετηθεί είναι διαθέσιμα. Υπάρχουν σχόλια. Όχι. Θεωρείται λοιπόν ότι εγκρίνονται τα πρακτικά και μπορούμε τώρα να περάσουμε στο πρώτο σημείο που ανακοίνωσα ήδη. Δύο λεπτά να ελέγξω και τα έγγραφα των 53 εκθέσεων. Να ζητήσω τώρα από την κυρία Γιάλα Σέντερ να πάρει το λόγο για τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω τον Πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου, τον κύριο Λένε. Επίσης χαιρετίζω ότι έχουμε εδώ και την Προεδρία του Συμβουλίου και τον κύριο Έτιγκερ. Καταρχήν, Βρισκόμαστε εν ώψη της τελευταίας απαλλαγής αυτής της θητείας. Πρόκειται για την απαλλαγή για το 2017 είναι ένα σημαντικό έτος για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός, αλλά αφετέρου είναι σημαντική και αυτή τη στιγμή το 2019 γιατί είμαστε μπροστά σε έναν απολογισμό και ακριβώς οι, οι νέες ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου θα είναι κλειδί για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε μία σύντομη αποτίμηση όλων αυτών ε, των ετών, 15 στην περίπτωσή μου, όπου μάθαμε από κοινού όλα τα θεσμικά όργανα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με κάθετο τρόπο με σταθερό τρόπο αλλά και με ανοιχτό πνεύμα προς τα άλλα θεσμικά όργανα έδρασε για να βρει τους καλύτερους δυνατούς ε, τρόπους και οδούς έτσι ώστε ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωσης να εφαρμοστεί εκεί όπου είχε αποφασιστεί, δηλαδή σε σχέση με τις προτεραιότητες και του στόχους. Και επίσης ε, να υπάρχουν και οι εγγύσει κανονικότητας και νομιμότητας. Πρέπει να σα ευχαριστήσω κύριε Λένε γιατί εκπροσωπείτε εδώ το Ελεκτικό Συνέδριο για την αξιοσημείωτη βοήθεια. Ήταν ε, πάρα πολύ σημαντική και το γεγονό ε, ότι είμαστε στο δεύτερο έτος που δεν είναι αρνητική δήλωση αξιοπιστίας και ανοίγει δυνατότητες μιας διαδρομής ε, βάσει της οποίας θα πούμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι άξιζε όλη αυτή η δουλειά τον κόπο, γιατί σε όλη αυτή την περίοδο μπορέσαμε να μειώσουμε σημαντικά τα ποσοστά λάθους, τα επίπεδα λάθους. Όμως είναι σημαντικό και το είπε και το Ελληνικό Συνέδριο και το συζητήσαμε και με την Κομισιόν εις βάθος, είναι απαραίτητο το εξή. Υπάρχουν νέε προκλήσει που εμφανίζονται. Παραδείγματο χάρη, όλο το θέμα των χρηματοοικονομικών μέσων που διαφέρουν πάρα πολύ και τα νέα τα ταμεία εμφανίζονται σαν δυνατότητα στον ορίζοντα. Ή επίση και το θέμα των δημόσιων εγωνισμών ή τα ε, διάφορα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την άμυνα, την κλιματική αλλαγή ή άλλες θεμελιώδεις πτυχές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά απαιτούν τη σοφία μας για το μέλλον. Το 2017 ε, προσπαθήσαμε για το 2017 να έχουμε μια ευανάγνωστη έκθεση έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να διαβάσουν ε, τι προχώρησε και πού έγκυται τα κύρια προβλήματα και προκλήσεις. Εργαστήκαμε για την άμεση διαχείριση, υπάρχουν κάποια ερωτηματικά που πρέπει να επιλύσει η Κομισιόν. Επίσης, εργαστήκαμε και στην ε, επιμερισμένη διαχείριση. Εκεί υπήρξε σημαντική βελτίωση. Σιγά σιγά ξεπεράστηκαν κάποια από τα κύρια προβλήματα και επίση και στην έμεση διαχείριση εργαστήκαμε όπου μέσω των ταμείων ε, και των οργανισμών χρειάζεται να πάμε πιο πέρα. Πέρα από το θέμα δηλαδή του ελέγχου του προπολογισμού. Στην ε, ψηφοφορία στην Επιτροπή και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους, τη Γραμματεία, και τι γραμματείε των ομάδων που μα βοήθησαν πάρα πολύ, συνέβησαν δύο νέα τεινά. Το ένα έχει να κάνει με την ε, κακή χρήση της ε, Όλαφ ε, σε σχέση με την οργάνωση EMG, τον οργανισμό EMG και επίσης κάτι άλλο που είχε να κάνει με την σύγκρουση συμφερόντων για το Γενικό Γραμματέα της Κομισιόν. Και φυσικά θα έχουμε τη συζήτηση και εγώ θα σας απαντήσω σχετικά στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Βάλη να πάρει το λόγο για 4 λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές για τη συνεργασία, την Επιτροπή, την, το λέκτικό Συνέδριο και την ΠΕΙ, την Τράπεζα Επενδύσεων για τα στοιχεία. Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προωθήσει την ανάπτυξη της χώρες είναι πολύ σημαντική. Επομένως, ε, ακόμη και ε, το, είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουμε τα σχετικά νούμερα. Θα αναφερθώ σε ένα από τα πιο σημαντικά θέματα. Το ελεκτικό συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του είπε ότι το ποσοστό λάθος για τις πληρωμές που έλαβαν χώρα το 2017 φτάνει στο 4,5%. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό στοιχείο και το υπογραμμίσαμε στην έκθεση. Οι πράξει όπου βρήκαμε τα περισσότερα λάθη σχετίζονται με τα ε, προγράμματα των επιδοτήσεων στι συμφωνίε τη εισφορά φοράς με του διεθνεί οργανισμού και με τις ε, οργανισμούς συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Η Κομισιόν θέλει να βελτιώσει τη δικασία των συμβάσεων και τη διαχείριση ε, των διαγωνισμών. Η DGDEFCO πρέπει να βελτιώσει τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικτών κλειδί για τα αποτελέσματα αποτελέσματα και τις επιδόσεις, συλλέγοντας ξεκάθαρες και πλήρες πληροφορίες. Θέλω να υπενθυμίσω ότι το 2017 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης δόθηκαν περίπου 860 εκατομμύρια ευρώ μέσω ε, της διαδικασίας στήριξης στον προπολογισμό. Υπάρχει σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη των χωρών που εποφελούνται από αυτό το μέσο και αυτός ε, ο τρόπος βοήθειας θα πρέπει να μεταμορφωθεί συγκεκριμένε δράσεις για να καταπολεμηθεί η απάτη. Υπάρχει υψηλό κίνδυνο εδώ. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε διάφορα επεισόδια φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή και παράνομων ε, χρηματοοικονομικών ροών, όπω ε, αναφερθήκαμε και στην έκθεση που ψηφίστηκε σήμερα. Θα ήθελα να αναφερθώ στα Trust Fund τη Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη μέχρι τώρα έχει συνεισφέρει περίπου 3 σε 4 συνολικά. Τα τα ταμεία είναι χρήσιμα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε κρίσιμε περιπτώσει, ε, όμω, χρειάζονται αυστηρό έλεγχο είτε στην, ε, προς τον προσδιορισμό των στόχων είτε στην υλοποίησή του. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να αυξήσουμε την εχνηλασιμότητα ε, των δράσεων και τη συνεργασία με τη ΜΚΟ και με του διεθνείς οργανισμού. Η συνεργασία είναι σημαντική, αλλά υπενθυμίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν αυστηροί μηχανισμοί ελέγχου και ακριβή. Υπενθυμίζω, το Ελεκτικό Συνέδριο πρόσφατα δημοσίευσε μια ειδική έκθεση για να αναλύσει την ανεχνευσιμότητα τη χρηματοδότηση τη Ένωση ε, για, ε, για κονδύλια που αφορούσαν τη ΜΚΟ. Υπογραμμίστηκε ότι η Κομισιόν δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική και βρέθηκαν ε, σημεία αδυναμία στη διαδικασία διαχείριση, αλλά και στη συλλογή πληροφοριών σε σχέση με τι υπεργολαβίε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ευχαριστήσω επίση του και το Ελεκτικό Συνέδριο, ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Σμίτ, επίση για τέσσερα λεπτά. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ κυρίε και κύριοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2017 δαπάνησε 1,9 δις ευρώ. Το ποσοστό σφαλμάτων ήταν πολύ χαμηλό, αλλά εν πάση περιπτώσει 0,4%. Ε, παρόλα αυτά το 0 βεβαίω θα ήταν ε, το καλύτερο. Τους ε, τελευταίους μήνες ε, προσπάθησα εγώ προσωπικά να εξετάσω όλους τους ομίλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι συνάδελφοι ήταν πολύ ειλικρινείς και βοηθητικοί. Μου έθεσαν στη διάθεσή μου όλα τα στοιχεία που γνώριζαν και είχα την αίσθηση ότι πραγματικά μου έδωσαν απολύτω ειλικρινεί απαντήσει. Βεβαίω, ό,τι λάβει δεν είναι χρυσό και βεβαίω στου τομεί από του οποίου προέρχονται τα περισσότερα παράπονα των συναδέλφων και εδώ είναι η διατροφή, τα κτίρια κλπ. Εδώ υπάρχει η ανάγκη να βελτιωθεί η κατάσταση. Παράδειγμα, η οδηγή ε, των των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Ε, έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις. Όπως σας είπα, ε, εξέτασε όλους τους τομείς, ε, η αξιωματούχοι σύνδεσης και με αυτό το θέμα ασχολήθηκα. Εγώ θεωρώ ότι οι σταθερές δαπάνες για τα κτίρια και τις δαπάνες είναι δυσανάλογα σε σχέση με τις δαπάνες για τους αξιωματούχους σύνδεσης. Και θα ήταν ε, προτιμότερο να είναι το έργο τους πιο αποτελεσματικό και θα ήθελα να υπάρξει στενότερη επικοινωνία με τα κοινωνικά μέσα. Δεν είναι αρκετό να ε, παίρνουν το λόγο μόνο όταν γίνονται κάποιες αρνητικές εκστρατείες, αλλά θα πρέπει να φροντίζουν να μην υπάρχουν καθόλου fake news. Επίσης, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους με την ευκαιρία αυτή ε, υπάρχουν ε, νέες... Ε, η συνεργασία ήταν πολύ επικοδημητική και το βλέπουμε στο αποτέλεσμα σχέση με τους συμβιβασμούς που επιτεύχθηκαν. Η πιο προβληματική τομής είναι το συνταξιοδοτικό ταμείο το βλέπουμε κάθε χρόνο. Εδώ ε, χρειάστηκε να βάλουμε το μυαλό μας να λειτουργήσει, γιατί οι λύσεις θα μπορούσαν να βρεθούν, γιατί και οι καιροί έχουν αλλάξει. Θα πρέπει να βρεθούν κάποιες ε, λύσεις, ούτως ώστε ε, πραγματικά οι βουλευτές οι οποίοι έχουν πληρώσει τις φορές τους να μπορούν να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους. Ε, τώρα, όσον αφορά την έδρα στο Στρασβούργο, ε, οι Γάλλοι συνάδελφοι δεν δείχνουν εδώ καμία κατανόηση, δεν θέλουν να γίνει καθόλου συζήτηση, αλλά θα ήθελα εδώ να σας υπεσημάνω τις δαπάνες ε, πάνω από 21 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος. Ε, είναι το κόστος αυτό. Τρίτον, το φάπαξ ποσό ε, έστω και αν έχει κανείς αντίθετη γνώμη θα πρέπει να το αποδεχτούμε. Ε, δεν είναι δυνατόν ε, να κάνουμε εδώ ατέρμονες συζητήσεις. Συνολικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι έγινε καλή δουλειά εδώ και ελπίζω να χορηγηθεί απαλλαγή στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Κόν επίσης για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Ελένε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το 2017 η εκτέλεση του προπολογισμού ήταν ικανοποιητική. Ε, διαπιστώθηκαν μόνο λίγες ατασταλίες και πέραν τούτου ασχοληθήκαμε με ειδικέ πτυχές της ε, διοίκησης και της διαχείρισης του προσωπικού. Ως εισηγητής ε, μου ήταν σημαντικό να εξασφαλίσουμε μια ισότητα για τις γυναίκες και να μην υπάρχουν φαινόμενα παρενόχληση στον χώρο εργασία. Και χαιρετίζονται πολλέ συστάσει του Κοινοβουλίου από την τελευταία απαλλαγή. Έχουν εδώ ληφθεί υπόψη και μπορούν να αξιολογηθούν ω θετική εξέλιξη όσον αφορά τη χρήση των πόρων στο επίπεδο τη διοίκηση και τη διαχείριση του προσωπικού. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, για παράδειγμα, έκανε κάποιε ε, προόδου ε, για παράδειγμα όσον αφορά την ε, προκήρυξη διαγωνισμού μέσω προχωρημένων συστημάτων πληροφορικής, κατάρτισης κλπ. Η, η Επιτροπή των Περιφερειών ε, επέδειξαν εξαίρετη διαχείριση και η μερασία των ε, κτηρίων και των υπηρεσιών οδήγησαν σε εξοικονόμηση. Ε, ωστόσο, έγιναν τεράστιες επενδύσεις στον αφορά την πληροφορική και το αίτημα περικοπής ε, των ε, κονδυλίων εδώ ε, το συμμερίζουμε. Οι συνάδελφοι έκαναν πολλές προσπάθειες να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους. μπόρεσαν να γίνουν οικονομίες και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, συνέπεια των συστάσεων του Κοινοβουλίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατέβαλε σημαντικές προσπάσεις όσον αφορά την επιτάχυνση των εργασιών του. Έτσι, ε, θέσπισε ένα νέο σύστημα διαχείρισης ε, ο διπλασιασμός του αριθμού των ε, δικαστών και η αύξηση των ε, υποθέσεων, ωστόσο είναι ζητήματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ε, εκπονεί τις εκθέσεις και μας υποστηρίζει ενεργά στη χορήγηση της απαλλαγής. Η εργασία επικοινωνίας με τους πολίτες επίσης είναι εξαίρετη. Ε, και βεβαίως όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, είναι σημαντικές οι εξελίξεις. Παρόλα αυτά υπάρχουν και ορισμένες, ορισμένα προβλήματα. Το Συμβούλιο δεν αναγνωρίζει το αίτημα απαλλαγής του Κοινοβουλίου. Προσπαθούμε να επεξεργαστούμε μια νέα συνεννόηση με το Συμβούλιο. Γι' αυτό θα ήθελα να συστήσω την αναβολή της απαλλαγής με την ελπίδα να σημειωθούν πρόοδοι στο μέλλον. Στην Επιτροπή Περιφερειών ε, ε, έχουν αποκαλυφθεί κάποιες ε, ατασταλίες ε, που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο συνάδελφο. Ε, με τον κύριο Κλίνξ ε, είπαμε ότι θα μπορεί να κινηθεί μια διαδικασία συνδιαλλαγής η οποία ελπίζουμε να οδηγήσει ένα καλό αποτέλεσμα. Στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υπήρξαν ε, ορισμένες, ορισμένα, ορισμένες παρατυπίες. Οι αποφάσεις βεβαίως για την κάθε επιμέρους περίπτωση θα πρέπει να γίνουν μέσω του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή. Η σοσιαλιστική πολιτική ομάδα έχει μηδενική ανοχή σε περιστατικά παρενόχλησης των γυναικών. Ε, επίσης σημειώθηκαν παρατυπίες όσον αφορά τις δαπάνες ταξιδίου και εδώ θα πρέπει να γίνουν βελτιώσεις στους κανόνες και θα πρέπει να καταχωρείται πιο αυστηρά η υποχρέωση παρουσίας των συναδέλφων. Υπάρχει πίεση χρόνου, επειδή έχουμε ψηφοφορία στις 5. Παρακαλώ λοιπόν να τηρείτε το χρονικό περιθώριο που σας δίνεται. Η κυρία Σαραβαμά για τέσσερα λεπτά επίσης. Ο κύριος Σαραβαμά, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε του Ορεντικού Συνεδρίου, κύριε Λένερ, κύριε Επίτροπε Έτιγκερ, κύριε Τσαμπάν, εξ του Συμβουλίου, αξιότιμα μέλη. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Οργανισμών και το επαλληλικό προσωπικό συμπεριλαμβανομένες της Γραμματείας και των επιτελείων μας, για την πολύ σημαντική δουλειά που έκαναν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απαλλαγής 2017. Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα προβεβλημένες σε επίπεδο κρατών μελών και επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Γι' αυτό και χαιρετίζουμε τα συνολικά θετικά αποτελέσματα ε, τη γνώμη ε, ε, και των ελέγχων μάλλον του Ελεκτικού Συνεδρίου για τη χρηματοδότηση αυτών των υπηρεσιών για αυτό το οικονομικό έτος. Υπάρχει λοιπόν γνωμοδότηση χωρί επιφύλαξη ό,τι αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και ό,τι αφορά την κανονικότητα και νομιμότητα των πληρωμών που προκύπτουν από του λογαριασμού αυτού για όλε τι υπηρεσίε για το 2017. Πλην των πληρωμών για το ΕΑΣΟ, για το σύστημα, ε, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης Ασύλου. Τα ζητήματα που οδήγησαν το Ελληνικό Συνέδριο να εκδώσουν αρνητική γνώμη ήταν, αφορούσαν βασικά την μη συμμόρφωση των αφορά πληρωμές ε, σε σχέση με τις ε, δημόσιες συμβάσεις. Όμω, εμείς ε, χαιρετίζουμε τις προθέσεις ε, για φιλόδοξε μεταρρυθμίσει, ε, και θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ανάπτυξη μια καλύτερης, πιο διαφανούς και αξιόπιστης δομή διακυβέρνηση. Γι' αυτό προτείνουμε να δοθεί η απαλλαγή σε όλες τις υπηρεσίες πλην του ΕΑΖΟ για το οποίο προτείνεται η αναβολή της ε, εκαθάρισης, της απαλλαγής. Θα ήθελα να κάνω τις εξής οχτώ οριζόντες παρατηρήσεις. Πρώτον, καλούμε τα, τις υπηρεσίες να συνεχίσουν να εφαρμόζουν ε, την, ε, τον καθορισμό του προβλογισμού με βάση τις επιδόσεις και να έχουμε αυτά αποτελέσματα και, από, και την απόδοση για να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να έχουμε προσθεθέμενη αξία. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το δίκτυο και οι επιμέρου υπηρεσίε θα πρέπει να εργαστούν από κοινού και να υπάρχει επικοδομητική ανατροφοδότηση, feedback καθ' όλη τη διάρκεια του ΠΔΠ και να διερευνώνται νέοι τρόποι χρηματοδότηση για του οργανισμού και τι υπηρεσίε. Τρίτον, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει έναν σωστό ε, τύπο για, την, ε, για τα συνεχιζόμενα έργα, τα carryovers και την διαμόρφωση του προλογισμού. Τέταρτον, καλούμε την Επιτροπή για τα, στα επόμενα έτη αυτομάτως να δίνει ε, τον απαραίτητο προπολογισμό και τα μέλη ε, του προσωπικού σε ό,τι αφορά τους 32 αποκεντρωμένους φορείς. Πέμπτον, μας προβληματίζουν ο αριθμός των ε, παραγόντων και οι αδυναμίες που εντοπίζονται στις δημόσιες συμβάσεις. Η νέα προσέγγιση που περιλαμβάνει και ιδιωτικούς φορείς οδηγεί σε σημαντική αύξηση του διοικητικού άχθους για τις υπηρεσίες. 7. Οι υπηρεσίε θα πρέπει να συνεχίσουν το σημαντικό του ρόλο σε ό,τι αφορά την αποτροπή συγκρούσεων ε, συμφερόντων, ε, των whistleblowers και του καθεξής. Και τέλος, πρέπει να δίδεται η απαλλαγή για το έτος νη συνένα, το επόμενο έτος δηλαδή από τη χρονιά για το οποίο δίνεται η απαλλαγή. Και χαίρομαι που έχει τεθεί στο, στη μέσα διάταξη το μεσημέρι και όχι βράδυ όπως γίνεται πάντα. Ευχαριστούμε. Κυρία Νταλμπάλοβα, για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κυρίε και κύριοι. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω του συναδέλφου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαίρομαι που καταφέρνουμε τώρα να αξιολογήσουμε ακριβώς το δημοσιονομικό έτος του 2017 και από οικονομική άποψη και από, πραγματικά, από πλευράς πραγματικού αντικτύπου. Εκτιμώ ιδιαίτερως ε, τη συνεργασία μας. Η αξιολόγηση ε, των επιδόσεων και των αποτελεσμάτων αυτών των κοινών ε, επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντική διαδικασία. σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του προλογισμού, αλλά και σε ό,τι αφορά ε, την ε, ενεργοποίηση και μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Ο συνολικός προπολογισμό ήταν 2,1 δις ευρώ το 2017, 2% του συνολικού προπολογισμού, με προσωπικό 700 άτομα, με στόχο ε, την έρευνα για την καινοτομία, για την αύξηση της τη της βιομηχανία ε, και την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων. Ε, επομένως, αυτές οι κοινέ πρωτοβουλίε είναι πολύ σημαντικές για να δημιουργηθούν μακρόπνοα προγράμματα σε αυτόν τον τομέα. Επομένω, η χρήση των κοινών επιχειρήσεων είναι ένα πολύ σημαντικό ε, μοχλό ανάπτυξη, γιατί διασυνδέει και τα ευρωπαϊκά κονδύλια αλλά και τα ιδιωτικά κεφάλαια. Και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποτελέσει έναν πιο σημαντικό φορέα στον τομέα τη έρευνα και καινοτομία. Πολύ σημαντικό εδώ είναι η εμπλοκή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Χαίρομαι που οι κοινέ επιχειρήσει υποστηρίζουν τι μικρομεσαίες ε, επιχειρήσει και ελπίζουν να αυξηθεί ε, η συμμετοχή του στο μέλλον. Το σημαντικό εδώ είναι ότι ο ορίζον 2020 συμπεριλαμβάνει και τους Key Performance Indicators, τους βασικούς δείκτες επιδόσεων. Και συγχαίρω τις κοινέ αυτές επιχειρήσεις, γιατί οι περισσότερες το 2017 είτε ε, επέτυχαν του στόχου ή και τους ε, ξεπέρασαν. Η αποδοτικότητα αυτών των κοινών επιχειρήσεων αποδεικνύεται από το γεγονό ότι ε, το διοικητικό κόστο είναι κάτω από το 5% και δείχνει αυτό λοιπόν ότι είναι ε, πολύ αποτελεσματική από οικονομική άποψη αυτοί οι μηχανισμοί. Ήταν πολύ πιο σύντομες οι προθεσμίες σε ό,τι αφορά την εκταμείευση των κονδυλίων από τα προβλεπόμενα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι κάποιες ε, κοινέ επιχειρήσεις πέτυχαν 7 από τους 9 βασικούς στόχους milestones που είχαν προβλεφθεί για το 2017 και από το 32 που ήταν το σύνολο έχουν επιτευχθεί 30 αυτή τη στιγμή. Για το Excel σε ό,τι αφορά την νομιμότητα και κανονικότητα αποδεικνύεται όμως ε, είναι αποτέλεσμα των ε, προηγούμενων του Άρτεμις και Έρνια και αφορά προηγούμενα ε, προγράμματα της προηγούμενης πραγματικής περίοδου. Θεωρώ ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι τα πήγαν πολύ καλά και συγχαίρω τις κοινέ επιχειρήσεις για τα αποτελέσματά τους. Ε, υπό το φω και της ομόφωνης απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα ήθελα και η Ολομέλεια να ε, δώσει την απαλλαγή. Ευχαριστώ. Το Συμβούλιο, παρακαλώ, έχει το λόγο. Εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, συγγνώμη κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό θα μπορούσα να σας ζητήσω να μην κάνετε φασαρία για να μπορούμε να συνεχίσουμε, παρακαλώ. Είναι ιδιαίτερη η τιμή μου να συμμετέχω σήμερα σε αυτή τη συζήτηση για την εφαρμογή του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χρηματοοικονομικό έτος 2017 στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας απαλλαγής για τον προπολογισμό όπως ε, προβλέπεται στο άρθρο 319 τη Το Συμβούλιο δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην ε, διαδικασία της επαλλαγή. Είναι σημαντικό τα ευρωπαϊκά κονδύλια χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες ε, και οι δαπάνε να σέβονται τις αρχές του αυτού δημοσιονομικής διαχείρισης. στι 20 Φεβρουαρίου η συνάδελφό μου, Λουμινίτσα Ντομπέσκου, ε, η μόνιμη εκπρόσωπο της Ρουμανία Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσίασε στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού τη σύσταση του Συμβουλίου για τη χορήγηση απαλλαγή των Κομισιών. Η Ολομέλεια θα ψηφίσει σήμερα και πιστεύω ότι θα επιβεβαιώσουμε την ψήφο τη επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και θα χορηγηθεί η απαλλαγή στην Κομισιόν. Αφενό, το Συμβουλίο καλωσορίζει το γεγονός ότι για δεύτερη φορά στη σειρά το λεκτικό Συνέδριο ε, γνωμοδοτεί με επιφύλαξη για την ομότητα και κανονικότητα των πληρωμών. Επίση, καλωσορίζουμε τη σταδιακή μείωση του συνολικού εκτιμόμενου ποσοστού ελέγχου, όπω ανέφερε το Λεκτικό Συνέδριο τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη, το Συμβούλιο λυπάται ότι το συνολικό εκτιμόμενο ποσοστό λάθου για τι πληρωμέ του 2014 στο 2,4% είναι πάνω από το όριο του 2%. Το Συμβούλιο, επομένως, επαναλαμβάνει την επιθυμία του να υπάρξουν περαιτέρω βελτιώσεις στα στήματα ε, δημοσιονομικής διαχείρισης και στα εκτιμόμενα επίπεδα λάθους σε όλους τους τομείς πολιτικής. Κυρίε και κύριοι, το έτος 2017 ήταν ιδιαίτερο όχι μόνο επειδή βρισκόμαστε στο μέσο της περίοδου που καλύπτεται από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά και λόγω των αλλαγών στο ε, πλαίσιο του ελέγχου ε, και της ε, αξιοπιστίας. Το λεκτικό συνέδριο έχει εισαγάγει μια νέα προσέγγιση. Για πρώτη φορά έλεγξε τα πακέτα της αξιοπιστίας που έχουν υποβάλει τα κράτη-μέλη για την σημερινή τρέχουσα για την σημερινή προγραμματική περίοδο. Έχουμε παρατηρήσει μια ε, σταθερή βελτίωση στη διαχείριση του προπολογισμού τα τελευταία χρόνια. Το συνολικό ποσοστό λάθο για τι πληρωμές μειώθηκε το 2017 για τέταρτη συναπτή χρονιά. Τα κράτη-μέλη και κομισιόν μπορούσαν να βελτιώσουν τα συστήματα ελέγχου και διαχείριση. Θα πρέπει να συνεχίσουμε την καλή δουλειά. Φυσικά υπάρχει η δυνατότητα βελτίωση ε, ιδιαίτερα στις πληρωμές αποζημιώσεων που εξακολουθούμε να βρίσκουμε το μεγαλύτερο ποσοστό λάθους. Είναι ιδιαίτερα πολύπλοκοι ακόμη οι κανόνες και για τους δικαιούχους για να τους ακολουθήσουν και για τις αρχές να τους ελέγξουν ένα ε, ρυθμιστικό πλαίσιο, απλούστερο, πιο διαφανές, θα είναι ουσιαστικό για να έχουμε αποτελεσματικό και σωστό έλεγχο των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το Συμβούλιο επίση μειώνει τη σύσταση του συνεδρίου σε ό,τι αφορά την απλούστευση και τον εξορθολογισμό των στρατηγικών πλαισίων που διέπουν την εφαρμογή του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Επίση, ε, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι ο προπολογισμό θα παρουσιάζει αποτελέσματα σε σχέση με του στόχου τη Ένωση. Οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι θα πρέπει να δουν ότι τα χρήματά τους ε, δεν ε, ξοδεύονται δεν σπαταλώνται, αλλά δαπανώνται σε ό,τι κάνει διαφορά και είναι σημαντικό για αυτούς. Γι' αυτό το Συμβούλιο υποστηρίζει τη σύσταση του Συνεδρίου για τον εξορθολογισμό των δικτών, για τις επιδόσεις του προπολογισμού και τη βελτίωση του εξορθολογισμού μεταξύ των γενικών στόχων και των ειδικών στόχων του προπολογισμού. Επομένως, να ενισχύσουμε τη λογοδοσία για τα αποτελέσματα και να αυξήσουμε τη σαφήνεια και τη διαφάνεια για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η αύξηση της εστίασης ε, στην μέτρηση των επιδόσεων, όμως δεν θα πρέπει να εμποδίσει το συνέδριο να συνεχίσει την ουσιαστική δουλειά του για τι αιτήσιε εκθέσει και για την παροχή εκτιμόμενα επιπέδων λαθών για όλου του τομεί ε, δαπανών για το σημερινό και το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στους τομείς 3 ε, και 4, όπου έχουμε αυξανόμενη πολιτική σημασία. Το Συμβούλιο βρήκε κάποια σημαντικά σημεία ανησυχία ε, σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό. Υπάρξει σημαντικό επίπεδο ε, κρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων και ο προπολογισμό αναμένεται επίση να έχει ενδεχόμενε υποχρεώσει. Το Συμβούλιο θα ήθελε η Κομισιό να βελτιώσει τι εκτιμήσει τη πληρωμέ και να ακολουθήσει τι σύσταση του συνεδρίου, να δώσει περισσότερε πληροφορίε για την κατάσταση ε, των υποχρεώσεων και τη χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων. Αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε την διαφάνεια και την προβλεψιμότητα τη χρηματοδότηση τη Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο φαίνεται να συμμερίζονται την ίδια προσέγγιση. Καλωσορίζουμε τι βελτιώσει να τις δουν όλοι και θέλουμε να δούμε την καλή δουλειά των κρατών μελών, της Κομισιόν και του Ελεκτικού Συνεδρίου να βελτιωθούν περαιτέρω. Πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στους Ευρωπαίους πολίτες και στους φορολογούμενους ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια χρησιμοποιούνται με έναν τρόπο υπεύθυνο και υπάρχει και λογοδοσία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα, φτάνω τώρα στον Επίτροπο Έτιγκερ. Παρακαλώ, εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχετε το λόγο. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι συγητέ και βουλευτέ. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Πρόεδρε του Συμβουλίου, αξιότιμε κυρίε και κύριοι. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την επικοδομητική διαδικασία χορήγησης απαλλαγή. Την κυρία Γιάλα Σάντερ, και του συναδέλφου της από την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Θεωρώ το σχέδιο έκθεσης πραγματικά πολύ αξιοσημείωτο επί της ουσίας και ε, ε, ικανό. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο ε, είναι, λειτουργεί ως μόνιμος πάροχος συμβουλών, τις οποίες συμβουλές συχνά ε, συνήθως ακολουθούμε και ε, το οποίο αξιολόγησε θετικά την εργασία μας. Για το έτος προϋπολογισμού 2007 εξετάσαμε, ε, το έτος 2017 είναι το τελευταίο έτος αυτής της ιδέας πριν από τις ευρωεκλογέ. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών και την Πρόεδρο κυρία Γκρέσλε για, την, ε, ε, για το εξαίρετο έργο της και το ζήλο που έχει επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Επιτρέψτε μου μετά από αυτά τα πέντε έτη να κάνω ένα σύντομο απολογισμό. Τα τελευταία χρόνια βελτιώσαμε σημαντικά την εκτέλεση του προπολογισμού επιχειρησιακά η, η Επιτροπή αλλά και από στρατηγική άποψη το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έβαλε τις επιδόσεις στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του. Προσπαθήσαμε με τα ισχνά μας μέσα να εκπληρώσουμε τις κοινέ μας προτεραιότητες και να δημιουργήσουμε μια προσθέμενη αξία. Η προσθέμενη αξία θα αποτελέσει το έμβλημα και για τις, τα επόμενα πολιτή δημοσιονομικά πλαίσια. Προσπαθήσαμε να προσθέσουμε τις διατάξεις και επίσης προσπαθήσαμε να εποφελθούν όλοι οι τελικοί δικαιούχοι με την χρήση, με την δυνατότητα χρησιμοποίησης κάποιων ε, λύσεων απλούστευσης του κόστους. Η κυρία Γκρέσλε μας βοήθησε σημαντικά στις διαβουλεύσεις και αυτή ήταν η αφετηρία για απλουστευμένα, ε, θα είναι μάλλον η αφετηρία για απλουστευμένες διαδικασίες στα επόμενα πολιτή δημοσιονομικά ε, προγράμματα μπορέσαμε να μειώσουμε το ποσοστό σαλμάτων ε, κατά το ίμιση, 2,4% και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας σε αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε να εξυπηρετήσουμε και τα, τους φορολογούμενους. Επίσης, αυξήσαμε την προστασία του προϋπολογισμού και δημιουργήσαμε ένα πλαίσιο για πρόληψη και για διορθώσεις. Ε, ε βελτιώσαμε συστήματα ε, διενέργειας των ε, ελέγχων και για στο πίπεδο των χωρών μελών, ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία τους ως βάση για τη δική μας εργασία. Το ελεγκτικό συνέδριο ε, δεν εξέδωσε αρνητική απόφαση, αλλά μια θετική απόφαση με κάποιους περιορισμούς, όπως έκανε και στο παρελθόν. Ε, η εκτίμησή του αφορά την ε, εκτέλεση του προπολογισμού ε, σε σχέση και με τα διάφορα επιμέρους προγράμματα. Οι απαιτήσει και οι συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου έχουν συμπεριληφθεί στις προτάσεις της Κομισιόν για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, ούτως ώστε τα χρήματα φορολογουμένων να χρησιμοποιούνται λογικά, με σόφρονα τρόπο και να δημιουργείται μια προσθέμενη αξία. Ε, η, η προσεχή διαπραγματεύση για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο θα αποτελέσει ένα συγκεκριμένο βήμα προ την κατεύθυνση αυτή. Οι ε, εκθέσει κυρίε και κύριοι δείχνουν μια ξεκάθαρη εικόνα για τι θετικέ εξελίξει στην εκτέλεση προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιθυμούμε να καταστήσουμε περισσότερο σαφές στον πολίτη ποια είναι η προστέμενη αξία για τον Ευρωπαίο πολίτη. Ο προπολογισμό είναι μικρός, αλλά είναι αποτελεσματικός. Επειδή δημιουργούμε μια προστατευμένη αξία, αποτελέσματα, τα οποία οι χώρες μέλη μεμονωμένα δεν θα μπορούσαν να πετύχουν, παρά μόνο με υψηλότερο κόστος ένα δίκτυο υποδομών, οδικός, σιδηροδρόμου για την ενέργεια, ε, για τις ψηφιακές υποδομές, ε, εργασία για τους ε, νέους, ενεργειακή ασφάλεια, ψηφιακή ιστορική αγορά, έρευνα, προώθηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλα, σε όλους αυτούς τους τομείς ε, προσπαθούμε, να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή ε, προσθέμενη αξία. Η έκθεση σας ε, κατονομάζει τομείς όπου, που επιδέχονται βελτιώσεις. Πρώτο κεντρικό σημείο αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Στην αρχή του 15 και 16 ε, υπήρξε χαμηλή απορρόφηση των κονδυλίων, η κατάσταση βελτιώθηκε το προηγούμενο χρόνο και αυτό το χρόνο ανέκτησε έναν, το ρυθμό ο οποίος είχε προγραμματιστεί. Και έτσι προβλέπουμε ότι εξελίξει το 2021-2022 εξελίξεις θα χαρακτηρίζονται από μια απλούσευση του δημοσιονομικού πλαισίου και θα υπάρξει αποδοτικότερη απορρόφηση. Δεύτερον, επιθυμούμε ε, τα ε, να είναι πιο αποδοτικοί. Ε, κάτι που το πετύχαμε και το επιβάλλουν και ο ΣΑ. Τρίτον, ε, ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα για τις επιδόσεις μας. Επίσης, το περιθώριο σφαλμάτων. Επιθυμούμε να πράξουμε ότι περνάει από το χέρι μας, ούτε ώστε το περιθώριο σφαλμάτων να μειωθεί περαιτέρω. Μετά από την εκτέλεση των προγραμμάτων και μετά από τη διενέργεια όλων των ελέγχων, έχουμε ένα απομείναν περιθώριο σφαλμάτων ε, του 2%. Ε, θέλουμε να το μειώσουμε περαιτέρω όπως σας είπα και θέλουμε να το έχουμε σαν ε, βάση των εργασιών μας. Τέταρτο σημείο, συγκρούσεις συμφερόντων. Θα ήθελα να δηλώσω στο Κοινοβούλιο με όλο το σεβασμό και αυτό ισχύει ειδικά για την Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών ότι η όξυση των διατάξεων σε σχέση με τη σύγκρουση συμφερόντων υποστηρίχθηκε από το Κοινοβούλιο, από την Ελόγω Επιτροπή. Και τώρα ε, παίρνουμε κάποια μέτρα, κάνουμε βήματα, ούτως ώστε να υποστηρίξουμε τις χώρες μέλη για τη διαμόρφωση διατάξεων περί σύγκρουση συμφερόντων ε, στο νέο κανονισμό ε, του προπολογισμού. Και θέλουμε επίσης να συνοδεύσουμε την διαδικασία διενέργειας ελέγχων εκ μέρους των χωρών μελών και έχουμε προγραμματίσει συναντήσεις με τους εκπροσώπους των χωρών μελών σε σχέση με βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της σύγκρουσης συμφερόντων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι, θερμά, προσκεκλημένο να συμβάλλει ενεργά σε αυτές τις συνεργασίες. Κυρίε και κύριοι, η Κομισιόν εξετάζει τις καταγγελίες σε σχέση με περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων στην Τσεχία. Ε, και θα ήθελα εδώ να σε επισημάνω ότι είναι σημαντικό να κάνουμε διάκριση μεταξύ ε, πράξεων που έγιναν πριν από τη θέση ισχύ του νέου κανονισμού ε, στις 2 Αυγούστου στο επίπεδο των χωρών μελών και μετέπειτα ε, περιστατικών μετά τη Δευτέρα Αυγούστου. Εμείς ε, βεβαίως θα εξετάσουμε και τις δύο χρονικές περιόδους, μετά την Δευτέρα Αυγούστου και πριν. Και στην ε, Γένοβα ξεκινήσαμε ένα σεμινάριο για την διενέργεια ελέγχων με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων. Και αυτοί οι εξωτερικοί έλεγχοι θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θέλουμε να εξετάσουμε κατά πόσο οι διατάξεις περί σύγκρουσης συμφερόντων έχουν τηρηθεί στο χρονικό διάστημα από το 12 έως το 2018. Όσον αφορά το επόμενο χρονικό διάστημα, παρακαλέσαμε τη τσεχική κυβέρνηση να μας πει ε, τι μέτρα έχουν ληφθεί προκειμένου να αποκλειστούν ευθύ εξ αρχή ε, περιστατικά σύγκρουση ε, συμφερόντων. Και αυτή τη στιγμή διενεργούμε ε, σχετικέ έρευνε σε σχέση με τα μέτρα που θέλει να λάβει η κυβέρνηση για να καταπολεμήσει τέτοια φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων. Ο Πρωθυπουργό μας διαβίβασε γραπτά ότι δεν ε, συμμετέχει ε, στις ε, λόγω διαδικασίες. Θα ήθελα να σας επενθυμίσω ότι η Κομισιόν την εποχή εκείνη δεν είχε προβεί σε πληρωμές από τα Ευρωπαϊκά Διαφορετικά και Επενδυτικά Ταμεία για προγράμματα της Αγροφερ στην ε, Τσεχία μέχρι ότου διευλευκανθεί πλήρως η κατάσταση στη χώρα αυτή. Οι τσεχικές αρχές έχουν αναμερθεί σχετικά ε, και, ε, και καλούνται να εξετάσουν την εγκυρότητα αυτών των στοιχείων. Είναι σημαντικό να επιδείξουμε μια συνέπεια αλλά και αντικειμενικότητα σε σχέση με μια ανάλυση των απαντήσεων και πάλι των τσεχικών αρχών σε σχέση με το ερώτημα κατά πόσο θα πρέπει να διορθωθούν κάποιες ε, δαπάνες. Σε κάθε έλεγχο της Κομισιόν ε, θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο έχουν τηρηθεί οι διατάξει όχι και εφόσον διαπιστώσουμε ότι δεν έχουν τηρηθεί θα λάβουμε μέτρα προστασίας του προπολογισμού και ε, διορθωτικά μέτρα και για το παρελθόν. Ε, και επίσης θα ενημερώσουμε σχετικά ε, το Κοινοβούλιο το εξαγγείλαμε το Δεκέμβριο του προηγουμένου έτους και τον, την, στην προσεχή ολομέλεια του Απριλίου θα συνομιλήσω μαζί σας ενδεχομένως ε, πριν τις εκλογές και στο τέλος του έτους θα, σας, θα αναφερθώ γραπτά στα θέματα αυτά. Όσον αφορά τους διορισμούς ψηλών αξιωματούχων τον περασμένο χρόνο που είναι επίσης αντικείμενο αυτής της έκθεσης θα μιλήσω μαζί σας τον προσεχή Σεπτέμβριο. Εκπρόσωποι των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μπόρεσαν να μας ε, αποδείξουν πώς, ε, ποιες, πώς πληρούν τις διαδικασίες αυτές και να μας παράσχουν ένα παράδειγμα βέλτιστων πρακτικών ο διορισμός του Γενικού Γραμματέα της Επιτροπής ε, είναι ένα θέμα ειδικού ενδιαφέροντος για σας στην έκθεση αυτή. Από το διορισμό του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει σε πολλές δηλώσεις, υπέβαλε, έθεσε πολλά ερωτήματα και από τον ε, Ombudsman. Ε, ε, προσπαθήσαμε στην Κομισιόν να απαντήσουμε εκτεταμένα διεξοδικά όλες τις ερωτήσεις και να επισέλθουμε σε όλα τα στοιχεία του φακέλου που έχουμε στη διάθεσή μας. Εγώ πιστεύω ότι ο διορισμός έγινε σε αρμονία με τον κανονισμό βάσει των ισχυσών διατάξεων. Ο Γενικός Γραμματέας ε, πληρεί το λειτουργήμα του σύμφωνα με τον κανονισμό. Ο πρόεδρος και όλοι οι επίτροποι έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Ο Γενικός Γραμματέας έχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα και την εμπειρία που είναι αναγκαία για την επιτέλεση του έργου του. Δεν έχουμε την πρόθεση να αναθεωρήσουμε την απόφασή μας και κάτι τέτοιο δεν είναι άλλωστε δυνατόν ε, όπως γιατί ε, όπως είπαμε τον Απρίλιο του περασμένου έτους ε, ένας ε, τέτοιος πιστοποιημένος ε, διορισμός δεν μπορεί να ανακληθεί. Ε, θα ήθελα να σας πω ότι η διαφάνεια και το δίκαιο είναι σημαντικά καθοριστικά, καθοριστικές αξίες για μένα και στο πνεύμα αυτό θα προτείνω σε υψηλά αισθάμενους ε, συναδέλφους να θέσουν υποψηφιότητα. Είμαι πεπισμένος ότι οι υψηλοί αξιωματούχοι της ε, Επιτροπής ε, θα πρέπει να αποτελούν ένα αξιόπιστο πλαίσιο για αυτές τις διαδικασίες. Στην περίπτωση στην οποία ανέφερε στην η κυρία Γιάλα Σέντερ, για το EMG. Ε, είχαμε συνεργαστεί στο παρελθόν σε σχέση με το EMG. Όπως ξέρετε από τις διαβουλεύσεις στην Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών η Κομισιόν εξέδωσε ένα κανονισμό για το... Ε, προσέβαλε μάλλον τον κανονισμό της EMG και ακολούθησε μια διατησία και το δικαστήριο δεν ακολούθησε την άποψη της Κομισιόν. Γι' αυτό εμείς θα προβούμε στις εκκρεμείς πληρωμές προς το EMG Κυρίες και κύριοι όλοι σας συμβάλλατε ενεργά και ε, συγκεκριμένα στην, κατάρτιση, στην εκτέλεση του προπολογισμού όσον αφορά την τήρηση των κανόνων και την καταπολέμηση της απάτης. Το σχέδιο έκθεση το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα έχει συγκεκριμένα αιτήματα ως αντικείμενο τα οποία εμείς ως Επιτροπή θα τα λάβουμε σοβαρά υπόψη μας και θα ενημερώσει την Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών ε, το φθινόπορο ε, σε σχέση με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Επιτροπή. Η εργασία σας ήταν πολύ επικοδομητική και θα οδηγήσει, θα καρποφορήσει. Φοβούμαι ότι αυτή είναι η τελευταία φορά να συζητήσουμε για την ε, απαλλαγή και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την ε, συναδελφική σας συνεργασία. Ευχαριστούμε πολύ τον Επίτροπο. Χαίρετε και τη ευγνωμοσύνη και εκτίμηση του Κοινοβουλίου. Κυρία Λένερ, έχετε και πάλι το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, αξιότιμοι κύριε Ότιγκερ αξιότιμοι εκπρόσωποι του, της Πρόεδρου Συμβουλίου, επειδή είναι το τέλος της ε, θητείας και είναι η τελευταία ευκαιρία για το Ελεγκτικό Συνέδριο να πάρει το λόγο, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους μας, ε, την Επιτροπή Ελέγχων των Προπολογισμών και συγκεκριμένα την κυρία Γκρέσλαν, ευχαριστήσω τον Επίτροπο κύριο Ότιγκερ, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και την Ομάδα Εργασίας για την εξαίρετη ε, συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια διάρκεια της συνολικής ε, θητείας και γι' αυτό το τελευταίο έτος εκτέλεση του προπολογισμού. Η, ε, η νομοθετική σας ε, δραστηριότητα αλλά και η δραστηριότητα ελέγχου του προπολογισμού στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων σας θεωρώ ότι και για τον Ευρωπαίο πολίτη είναι καθοριστικό να εφαρμόζεται σωστά η ευρωπαϊκή νομοθεσία και να αξιοποιούνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η διαδικασία χορήγησης ε, απαλλαγής δεν είναι μια επιταγή εν λευκό, αλλά είναι ένα απόσπασπο κομμάτι μιας μακράς διαδικασίας συνεργασίας. Από τις ε, συνθήκες προκύπτει το εξή. Η Ευρωπαϊκή είναι νομικά υποχρωμένη να λάβει όλα τα μέτρα ε, προκειμένου να συμπεριλάβει τι παρατηρήσει του Κοινοβουλίου και τι εξηγήσει του Συμβουλίου στη διαδικασία χορήγηση απαλλαγή. Πιστεύω ότι εντωμεταξύ είστε εξοικειωμένοι με τι διαπιστώσει τη ετήσια ε, έκθεση και τη ειδική έκθεση του 2017. Όπω και το 2016, ε, δώσαμε, εκδώσαμε μια απόφαση η οποία είναι θετική με κάποιου περιορισμού. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι το ποτήρι είναι κατ' γεμάτο και είναι επιβεβαίωση τη θετική εξέλιξη τον τρόπο με τον οποίο η Κομισιόν και οι χώρες μέλη ε, διαχειρίστηκαν τα ευρωπαϊκά οικονομικά. Ε, και θα ήθελα εδώ να σε επισημάνω περισσότερο τέσσερα σημεία. Όσον αφορά τον έλεγχο της οικονομικής ε, επίδεση, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που συμπεριέλαβε τι συστάσει του ελεγκτικού συνεδρίου. Αυτός είναι ένα τρόπος βελτίωση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι τα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου και το προσωπικό μας ε, ε, ε βρίσκεται στη διάθεσή και μετά την έκθεση της έκθεσής μας. Ε, μπορείτε να απευθύνετε σε εμά αν θέλετε διευκρινήσει επιπλέον πληροφορίες. Είμαστε εδώ προκειμένου να σας συνδράμουμε στο έργο σας ως κοινοβουλευτικούς. Δεύτερον, προς τα ΡΑΛ, τα υπόλοιπα προς ε, καθάριση, διαπιστώνουμε ότι το Κοινοβούλιο ε, συμμερίζεται τις ανησυχίες μας. Όταν το περασμένο Οκτώβριο ήμουν εδώ, σας υποσχέθηκα να εξετάσω περαιτέρω αυτή την προβληματική. Γι' αυτό χαίρομαι πολύ που πλέον ολοκληρώσαμε τη σχετική μας ανάλυση ε, και διαλευκάναμε πώς έχουν τα πράγματα με τα ΡΑΛ. Η ανάλυση αυτή θα δοθεί στη διάθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού σε μια κοινή συνεδρίαση στις 2 Απριλίου. Ε, τρίτον, το αίτημά σας για την ε, Επιτροπή να εκπονήσει μια μεθοδολογία για τον υπολογισμό των σφαλμάτων που να είναι συγκρίσιμο με αυτήν του ελεγκτικού συνεδρίου θα πρέπει να οδηγήσει σε μια συμφωνία μεταξύ των δύο οργάνων και επιτρέψατε μου να επαναλάβω ότι σε αυτό το σημείο συμφωνούμε απολύτω. και ανεξάρτητα από την ε, δική μας ανεξαρτησία βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες της Επιτροπής προκειμένου να εξετάσουμε μέχρι πότε μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ο κ. Ε, αργότερα θα τοποθετηθεί εδώ, αλλά επιτρέψατε μου ήδη τώρα να συγχαρώ τον ίδιο και την ομάδα για τις πρώτες θετικές επαφές στο ζήτημα αυτό. Ε, διαπιστώνουμε ε, την, ε, τις, ε, ε, αναμένουμε με ενδιαφέρον μάλλον τις πρόοδους που πρέπει να σημειωθούν τους προσεχείς μήνες και εβδομάδες. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να επισέλθω σε ορισμένα σημεία τα οποία, στα οποία αναφέρεται ο Συμβούλιο στις δικές του συστάσεις. Φυσικά είναι και ο δικός μας στόχος ή δυνατόν να έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό πληροφοριών και να στις παράσχουμε ιδιαίτερως όταν αφορά, όσον αφορά το κόστος. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, χρειαζόμαστε για την ετήσια μας έκθεση σχεδόν το ίμιση των πόρων μας. Αυτό είναι πολύ υψηλό ποσοστό. Και όσο περισσότερο κινούμεθα ε, προς το ε, προς την ε, βελτίωση της ανάλυσης ε, κινδύνου τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα. Τώρα, έχουμε κάνει μια ανάλυση όσον αφορά τους υψηλότερους κινδύνους και θέλουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να έχουμε λεπτομεριακές πληροφορίες και να επιβεβαιώσουμε και τις πληροφορίες άλλων αξιολογητών. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε οι πληροφορίες αυτές βεβαίως να είναι επαρκού ε, επίπεδο εξοπιστίας. Όσον αφορά το 2017, έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση για τον τομέα της συνοχή. Ε, καινοφανές είναι το στοιχείο ότι οι έλεγχοι των ελέγχων που είχαν διενεργηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες αυτή τη φορά επαναξιολογήθηκαν και συμπεριλήφθηκαν στη δική μας αξιολόγηση. Με αυτή τη νέα προσέγγιση θέλουμε να σας συνδράμουμε με περιεκτικές πληροφορίες για τη διαχείριση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την υπεύθυνη διαχείριση ε, και για την συμμετοχή σας, την υπεύθυνη διαχείριση της ε, ε, έκθεσης αυτής. Έχουμε σαν σκοπό να χρησιμοποιήσουμε την προσέγγιση αυτή σε όλους τους τομείς του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί όπου τα αποτελέσματα είναι αξιόπιστα. Τέταρτον, ε, μία παρατήρηση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία αναφέρεται και στο δικό σας ψήφισμα όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που χρειαζόμαστε για το έργο μας. Ε, μπορέσαμε να βελτιώσουμε τουλάχιστον ε, το κλίμα της συνεργασίας και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δείχνει ενδιαφέρον να συμμετάσχει σε ένα διοργανικό διάλογο για τη σύνταξη ενός ε, μνημονίου συνεργασίας, το οποίο εμείς τις αποστήλαμε και πιστεύω ότι αυτή η εξέλιξη ε, οφείλεται και στην δική σας υποστήριξη ε, θα πρέπει να γίνουν το ταχύτερο δυνατό τώρα όλε αυτέ οι συνομιλίε και να ολοκληρωθούν μέχρι τη θερινή παύση. Θα ήθελα ωστόσο να σα κάνω μια θερμή έκκληση να παρακολουθήσετε του σύνεγγυ αυτέ τι εξελίξει και ή δυνατόν στην προσεχή θητεία να αναλάβετε την νομοθετική σα δραστηριότητα σε περίπτωση που ο διάλογος με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει οδηγήσει στο ευκταίο αποτέλεσμα και ε, ε, επίσης να ασχοληθείτε με το θέμα του, της περιστολής ε, της δικής μας εντολής ε, στον τομέα εποπτείας των τραπεζών. Κυρίες και κύριοι, η προεκλογική εκστρατεία θα ξεκινήσει λίγες εβδομάδες τουλάχιστον σε 27 χώρες μέλη και ίσως είναι οι σημαντικότερες ευρωεκλογέ αυτού του τύπου αυτή τη φορά. Γι' αυτό θα ήθελα να πω σε όλους τους βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου να αξιοποιήσουν στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας ε, τη δική μας, ε, το, ε, τις δικές μας αμερόληπτες εκθέσεις και στοιχεία. το Φεβρουάριο αυτού του έτους συνοψίσαμε τις εργασίες μας σε σύντομες παρατηρήσεις και θα συμπελάβουμε τις σκέψεις αυτές στην εκπόνηση του προσεχούς πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ωστόσο, εκδώσαμε και πολλές ειδικέ ε, εκθέσεις με σημαντικά στοιχεία. Ως ελεγκτές ε, δεν έχουμε την προτεραιότητα να στυλιτεύσουμε ή να μεμφθούμε τα άλλα ε, όργανα, αλλά κυρίως να τα συνδράμουμε με μια ε, ε, με αξιόλογα στοιχεία. Έχουμε καθυστερήσει επειδή είχαμε τόσο εκτενείς ε, τοποθετήσεις, γι' αυτό και δεν θα επιδείξω καμία ανοχή σε ό,τι αφορά το χρόνο. Παρακαλώ λοιπόν να τηρείτε το χρόνο που σας έχει απονεμηθεί. Με κάθε σεβασμό δεν θα σας δώσω περισσότερο περιθώριο. Τώρα, Εξ ονόματο ε, τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, η κυρία Γκίλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, και χαίρομαι που βλέπω τον πρώην συνάδελφο, κύριο Ελένε. Τα συμπεράσματά μου σε ό,τι αφορά την